Okay. Uh, good afternoon everybody. Um, Καλησπέρα σας. Μου συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Συζητούσαμε λίγο τις διαδικασίες. Αλλά τώρα θα συζητήσουμε την προστασία των θυμάτων ε, εγκλήματος και όπως ξέρετε έχουμε μία κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και βεβαίω αυτό αποδίδει την σημασία αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδουν οι δύο επιτροπές στο θέμα αυτό και νομίζω πως είναι μια συνεισφορά στην ενίσχυση ε, της ε, προστασίας των μαρτύρων αλλά πριν δώσω τον λόγο στους ε, εισηγητές. Θα ήθελα να τονίσω ακόμη μια φορά την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο εισηγητών και των δύο επιτροπών. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Τον λόγο που τώρα οι ε, εισηγήτριες. Αποφασίστε ποιος ε, θα μιλήσει πρώτος. Κυρία Καμίνες, ούτως ή άλλως είναι και μαζί μου. Thanks. Nice. Uh, it was a pleasure. It's a pleasure for me to to co-share this important joint meeting. Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση για μένα να λαμβάνω το λόγο. Υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα και το είπα και στην Επιτροπή Λίμπε Έχουμε τη συνεδρίαση δύο επιτροπών ταυτόχρονα ε, με κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε δύο διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα μέσα στο Κοινοβούλιο. Είδω λοιπόν μόνο τρία, τρεις βουλευτές από την ΛΥΜΠΕ είναι εδώ μαζί μας. Εγώ δεν είμαι μέλος της ΛΥΜΠΕ βέβαια, αλλά γνωρίζω ότι η ΛΥΜΠΕ συνεδριάζει ε, μαζί με μια άλλη επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε εδώ και θα παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή. Είναι λυπηρό που δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί ε, όπως πρέπει. Διότι αφορά εκατομμύρια ανθρώπους και θα έπρεπε να επιδείξουμε μεγαλύτερο σεβασμό και προσοχή. I just wanted to express this and not ε, δεν επιρρύπτω την ευθύνη σε κανέναν, αλλά ήθελα να το πω αυτό για να ε, θέσω τα πράγματα στη θέση τους και συμφωνώ με τον κύριο Τζούση ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά μάλιστα και ελπίζω αυτό να το διαπιστώσετε στην έκθεση. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την Γραμματεία και τους συμβούλους και τους σκιώδεις συγητές και μάλιστα κάποιοι είναι εδώ μαζί μας. Να τους ευχαριστήσω λοιπόν όλους που μας βοήθησαν με τις απόψεις και τις νομοδοτήσεις τους. Και πιστεύω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Τώρα κάνουμε τη δεύτερη παρουσίαση ουσιαστικά και ήδη έχουμε το, είχαμε τον τέταρτο γύρο του τριμερούς διαλόγου εχθές. Σε στενή συνεργασία με τους κοιόδης προσπαθούμε να προωθήσουμε τα πιο σημαντικά θέματα που, για τα οποία έχουμε εντονή εντολή να προωθήσουμε, να αναζητήσουμε τη βέλτιστη δυνατή συμβιβαστική λύση. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν κάποια άρθρα επί των οποίων δουλεύουμε ακόμα και υπάρχουν ακόμα κάποια εκρεμή θέματα. Τα περισσότερα από τα άρθρα που λάβατε την περασμένη φορά έχουν ήδη διευθετηθεί το 1, 3, 25, 18, 17, 11. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι με το άρθρο 2 μέχρι στιγμής και κυρίως είναι το άρθρο με τους ορισμούς. Οι δύο ορισμοί για την βία επί τη βάση της διαφοράς φύλων και η, σχέση, η βία σε στενές σχέσεις δεν έχουν περιληφθεί στις προτάσεις του Συμβουλίου. Τα συζητήσαμε αυτά και κατά τη διαπραγμάτευση καταλήξαμε ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί εάν δεν έχουν όλα συμφωνηθεί. Και ζητήσαμε να ξαναφέρουν αυτούς τους δύο ορισμούς, δεδομένου ότι τους χρησιμοποιούμε στα άρθρα 8α, β, 21, 22, 23, 25 και στα εδάφια και δεν θα ήταν σωστό, δεν θα ήταν σωστή νομοθεσία να, εάν οι ορισμοί που χρησιμοποιεί εάν μάλλον χρησιμοποιεί όρους για τους οποίους δεν δίδεται ο σωστός ορισμός για να χρησιμοποιείται με την ίδια έννοια σε όλες τις χώρες μέλη. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τους ορισμούς για ευθύς εξ αρχής. Άρθρα 8 και 8α. Στη συνέχεια. Δικαίωμα πρόσβασης των θυμάτων σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το άρθρο 8 τώρα μιλά για το δικαίωμα πρόσβασης και το 8α είναι η βοήθεια που είναι στη διάθεση των θυμάτων. Όλα αυτά τα δικαιώματα έχουν γίνει αποδεκτά από το Συμβούλιο και τώρα δουλεύουμε στο 8α, πάνω στο 8α, που αν θυμάστε ε, αφορά στα προσωπικά χαρακτηριστικά της ε, αξιολόγησης του κάθε ατόμου για να αποφασιστεί τι είδους υποστήριξη θα προσφερθεί και τι είδους εξειδικευμένη υποστήριξη θα προσφερθεί. Ε, το Συμβούλιο δυστυχώς δεν δέχθηκε την ψυχολογική υποστήριξη και το σημείο C γάμα προβλέπει συναισθηματική υποστήριξη. Για μας δεν είναι σαφής αυτή η διατύπωση, διότι μπορεί να περιλαμβάνει ένα φάσμα ε, ενεργειών ή μη ενεργειών, δηλαδή από το να ενθαρρύνει έναν άνθρωπο μέχρι να του δίνει μια... να του δίνει... τον χαϊδεύει ας πούμε ή τίποτα ή να, προσφέρει... να μην προσφέρει τίποτα. Εδώ θα έπρεπε να εμπλέκονται εξειδικευμένα άτομα, ψυχολόγοι και ελπίσεις Θέλουμε να αλλάξει η θέση του Συμβουλίου που προβλέπει οι χώρες μέλη να προάγουν, να προαγάγουν κάποιες υπηρεσίες με την εξής διατύπωση. Να, για να αναπτύξουν και να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Εμείς ε, θέλουμε να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα. Ε, ε, το χάρη να υπάρχουν ειδικά ειδικοί χώροι, καταφύγια κατά κάποιο τρόπο, όπου θα προσφέρεται ιατρική βοήθεια για θύματα από ε, βία που προέρχεται ε, που είναι καρπός της διάκρισης των δύο φύλων ή από βία μεταξύ προσώπων που έχουν στενή οικογενειακή σχέση κλπ επί τη βάση των προτάσεων που έχει κάνει το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια έχουμε το άρθρο 21. Αυτό ε, δημιουργεί πρόβλημα, διότι υπάρχει η ατομική αξιολόγηση και υπάρχει ένας κατάλογος κριτηρίων για κάποιες ειδικέ κατηγορίες. Γενικώ λέμε κατηγορίες και κατάλογος. Το Συμβούλιο αποδέχθηκε τις κατηγορίες όχι, ε, δέχτηκε τον κατάλογο, λέει η ομιλήτρια, τον κατάλογο για την αξιολόγηση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί την μνήα των διαφόρων κατηγοριών θυμάτων, όπως ε, ε, θύματα τράφικινγκ, βίας εξαιτίας διαφοράς φύλου, σεξουαλική βία και εκμετάλλευση και βία εναντίον ατόμων με αναπηρίες. Τώρα, εμείς προτείνουμε ένα συμβαστικό κείμενο το οποίο αναφέρει ολόκληρο τον κατάλογο όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο, όλα τα κριτήρια, αλλά στο πλαίσιο της ατομικής αξιολόγησης τώρα συντάξαμε τρεις παραγράφους, επί των οποίων προτείνουμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή πρώτον σε ε, θύματα τα οποία υπέστησαν σοβαρή βλάβη εξαιτίας του, της βαρύτητας της βίας, επίσης θυμάτων από διακρίσεις εις βάρους τους και θύματα που εξαρτώνται από τον δράστη και για τις τρεις αυτές κατηγορίες θεωρούμε ότι αυτές και για τις τρεις, τις τρεις αυτές κατηγορίες λοιπόν τις αναφέρουμε ξεχωριστά όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο. Και έρχομαι τώρα στο άρθρο 22 που είναι ένα δευτερεύον θέμα και, και το Συμβούλιο παραδέχθηκε ότι πρόκειται για παράληψη. Είναι το δικαίωμα για, για τα θύματα να έχουν ειδική προστασία κατά τη διάρκεια της διδικαστικής διαδικασίας. Δηλαδή, τα θύματα σεξουαλικής βίας, βίας εξαιτίας του φύλου και ε, θύματα που είναι και άτομα με ειδικέ ανάγκες πρέπει να τύχουν ειδική προστασίας. Επίσης της βίας από στενή σχέση. Α, η βία μεταξύ ατόμων που έχουν στενή σχέση έχει παραλυφθεί αλλά είναι παράληψη μόνο και δεν είναι επί τούτου. Όπως είπα, έχουμε και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ίδια κατεύθυνση. Και υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που διατυπώθηκαν από χώρες μέλη, δηλαδή ε, σχετικά με τη βία επί τη βάση του φύλου και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Έχουμε την ισχυρή υποστήριξη όλων των σκιωδών, εισηγητών και υπάρχουν και ισχυρές εντολές τις οποίες όλοι εσείς στηρίζετε. Γι' αυτό και θα παρουσιάσουμε έτσι την πολύ στεναρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προχωρήσουμε σε δευτερεύοντες ε, συμβιβασμούς και μόνον. Ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω ισπανικά. Ναι, η εμπιστοσύνη στην ε, δικαιοσύνη είναι προτεραιότητα για όλους τους ε, πολίτες και κυρίως για τα θύματα και θα πρέπει να εγγυόμεθα τα δικαιώματά τους ε, και είναι διάφανη η δικαιοσύνη παντού σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό απαιτείται και μάλιστα επιγόντως Εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε στα προστάγματα στο Στοχόλμης θα πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα και των θυμάτων και της οικογένειάς τους, να τους υποστηρίζει και ταυτόχρονα να βοηθούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε ένα εθνικό σύστημα δικαιοσύνης και δίπλα τους ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια εναρμόνιση ελάχιστων προδιαγραφών και εμείς δίνουμε έτσι τη μάχη μας και όταν από το Συμβούλιο ε, βλέπουμε ότι ιδιαίτερα στηρίζει πράγματα στην εθνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συντάξουμε καλά αυτή την οδηγία και να βελτιώσουμε την εθνική νομοθεσία, να την αρμονίσουμε. Και εμείς έχουμε διάφορα σημεία όπως το δικαίωμα για τα ενημέρωση και για τη διερμηνία και τη μετάφραση, επίσης στήριξη για τους για τα θύματα, δικαίωμα για την προστασία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έρευνα για το έγκλημα που έχει διαπραχθεί. Και η οδηγία αυτή αντιμετωπίζει μια δύσκολη καμπή ένα τριμερής διάλογος, ιδιαίτερα ευρύς και που έχει προχωρήσει χάρη στις προσπάθειες της Δανικής Προεδρίας για μια συνένεση, μια συμφωνία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και την Επιτροπή που δίδυξε από την αρχή ότι υποστηρίζει το Κοινοβούλιο εδώ αλλά υπάρχει και ένα θεμελιώδης δικαίωμα ακριβώ για κάποιον που ενδεχόμενα είναι βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται να ισχύσει και το δικαίωμα για ενημέρωση, για στήριξη, μετάφραση και διερμηνία και επίσης να αλλάξει γνώμη αν δεν θέλει να προχωρήσει σε δικαστική δίωξη. Εδώ υπάρχουν πολλές χώρες όπου υπάρχουν διάφορα δικαιώματα όπως και έφεσης θα πρέπει να δούμε μια κάπως πιο προχωρημένη ρύθμιση. Και ακόμα θα πρέπει να δούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα ακριβώς των θυμάτων ε, που πρέπει να ε, δούμε τι ρόλο μπορούν να παίξουν αυτά τα θύματα στην όλη ποινική διαδικασία. Και η Συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Υπάρχουν βέβαια πολλά ε, ελάσσονα εγκλήματα όπου δεν έχουν σημασία αυτές οι λεπτομέρειες αλλά αυτό θα πρέπει να διορθωθεί σε μερικές φορές ε, που είναι ιδιαίτερα βαριά τα εγκλήματα. Μερικές φορές ε, τα θύματα δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αλλά πρέπει τα ίδια να το δηλώσουν. Πάντως επαναλαμβάνω χρειάζεται η μετάφραση, η διερμηνία ακόμα και όταν δεν συμμετέχουν στην ολυπηνική διαδικασία. Εδώ είναι τα 5, 7 και 10 άρθρα. Στο άρθρο 21 τώρα είναι μια έκθεση οριζόντια, δεν πρέπει να θεωρείται κανένα θύμα χαμηλότερο από το άλλο, λιγότερη σημασία από το άλλο. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι όταν μιλάμε για τον κατάλογο αυτό που νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα σε αρκετές χώρες όπως και σε αρκετά από τα μέλη μας που θα φανεί σε λίγο. Εμείς ε, σε καμιά στιγμή δεν θέλουμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στα θύματα. Ξέρουμε ότι το ίδιο σημαντικά είναι όλα τα θύματα. Υπάρχουν όμως και θύματα που μπορεί να είναι διπλά θύματα και μιας ε, τρομοκρατικής ενέργειας είτε στην οικογένεια και χρειάζεται την προστασία για να μην επιστρέψει στην οικογένεια. Θέλουμε να υπάρχει μια αναφορά σε αυτά τα παραδείγματα και θα μπορούσαμε αυτό να το συμφωνήσουμε και να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε μια σειρά παραδειγμάτων για αυτά τα θύματα και έτσι να συμπεριλαμβάνεται αυτή η αναφορά. Και μιλάμε ακόμα για την μεμονωμένη ε, αντιμετώπιση κάθε θύματος με ειδικέ περιπτώσεις και σε ειδικά σημεία. Βέβαια η κατάσταση αυτή είναι κάπως περίπλοκη, αλλά υπάρχουν και θύματα από τρομοκρατία που φοβούνται αντίπεινα, τα εκφοβίζουν οι εγκληματικοί, οι τρομοκρατικοί κύκλοι και ταυτόχρονα βέβαια και στην οικογένεια το ένα το άλλο. Χρειάζεται όμως όλα αυτά να τα γνωρίσει η κοινωνία και χρειάζονται περισσότερη προστασία σε μερικές περιπτώσεις και άλλα εγκλήματα με ειδικό, ιδιαίτερα ειδικό χαρακτήρα και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό όπως ε, ε, άτομα που δεν είναι κανά να μυθούν και τα παιδιά επίσης ε, που θα πρέπει αυτά να αναφερθούν ειδικά. Και ακόμα το άρθρο 27 που μιλάει για στατιστική στοιχείων, γιατί διαθέτει κάθε κράτο στοιχεία στατιστικής για τα εγκλήματα. Δεν μπορούμε να συγκριθούν. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε στοιχεία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Θέλουμε να ζητήσουμε την εφαρμογή ανάλογα με την εθνικότητα, την ηλικία, το φύλλο, όπως στην τροπολογία 24 έχουμε ζητήσει. Έχουμε ήδη τον αριθμό εγκλημάτων και θα ήθελαμε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή στοιχείων, πληροφοριών, να χαρακτηρίσει περισσότερο τις επαφές ανάμεσα στα διάφορα κράτη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δανική Προεδρία γιατί καταβάλε κάθε προσπάθεια για να συνταχθεί ένα καλό μέσο, ένα καλό εργαλείο και εμείς ε, προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τις απόψεις μας όπως είπαμε και προηγουμένως και πιστεύουμε ότι το θα μπορούσαν να λυθούν προβλήματα όπως αυτά που εντοπίζουμε και θέλουμε να προσφέρουμε ένα σωστό μέσο και εργαλείο τα θύματα, βελτιώνοντας την νομοθεσία και εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Στοκχόλμας να εγγυηθούμε την προστασία των θυμάτων στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε. Σύντομα, να πω το εξής. Δεν σας ενημερώσαμε για κάτι πολύ σημαντικό που αφορά το πακέτο των παιδιών Το πακέτο λοιπόν αυτό το είδαμε σε ένα πολύπλοκο ζήτημα και οι περισσότερες διατάξεις είναι κατά από την ομπρέλα των θυμάτων με συγκεκριμένες ανάγκες αλλά λάβαμε υπόψη και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα βέβαια υπήρξε η πρόταση της κυρίας Γκρίσμπεκ που υπάρχουν τώρα ως ε, ειδικέ διατάξεις που καλύπτουν τα παιδιά σε όλη αυτή την ομοθεσία Οτιδήποτε αφορά όχι μόνο τα παιδιά αλλά όλα τα θύματα είναι υπό την ε, ομπρέλα αυτή ε, στις συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα και με την ατομική αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πως είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για τη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι εξαιρετική δουλειά και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη για το ότι θα υπερασπιστείτε την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τις προσπάθειές σας, τις ώρες που αφιερώσατε. Τώρα, για την θέλει το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Κυρία Μπελάντα Τοντίνο. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, ήθελα μόνο να πω σύντομα πως πράγματι η Κομισιόν ε, στήριξε αυτή την έκθεση. Πολλές τροπολογίες σας είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα ε, δικαιώματα των θυμάτων και είμαστε ικανοποιημένες για το ότι έχουμε, έχουν καταφέρει τα κράτη-μέλη να κάνουν πολλά. Υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα, όπως ανέφερε η συγγήτρια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθεί μια καλή λύση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουμε ένα καλό κείμενο το οποίο πραγματικά θα δώσει ε, πραγματικά ρεαλιστικά δικαιώματα στα θύματα αλλά μην ξεχνάτε πως τα κράτη-μέλη πρέπει να τα εφαρμόσουν αυτά. Οπότε είναι λεπτή η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά είμαι σίγουρη πως θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γιάννη Σίντερτε από την Δανέζικη Προεδρία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξ της Προεδρίας να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας ε, προς τις δύο συγκήτριες για τη δουλειά που έχουν κάνει, που αντικατοπτρίζει το μεγάλο ενδιαφέρον των δύο επιτροπών για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στην Ευρώπη. Όπως ανέφεραν οι ε, οι έχουμε κάνει πολλή δουλειά για να βρούμε συμβαστικές λύσεις ε, στις θέσεις που ενδιαφέρουν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Έχουμε κάποια ζητήματα και σύμφωνα με τους υπολογισμού μας νομίζω πως μπορούμε να περιμένουμε κάποιον συμβασμό. Να ευχαριστήσω λοιπόν τις δύο εισηγήτριες για το ενδιαφέρον που έδειξαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι και οι δύο ικανές διαπραγματεύτριες αλλά παίζουν και επικοδομητικό ρόλο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους για να τους ακούσουμε. Πρώτα απ' όλα Κέρκοπ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τις συζητήτριες για την ε, δουλειά αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική και χαίρομαι για το ότι υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση της από το Συμβούλιο. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που αφορά και τα θύματα και τα εγκλήματα. Οι μεμονωμένες αξιολογήσεις για τα εγκλήματα και τα θύματα ε, απαιτούνται πάντα. Κανένα έγκλημα και κανένα θύμα δεν είναι ποτέ ακριβώς το ίδιο με ένα άλλο. Γι' αυτό θα έλεγα να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην μπούμε σε έναν κατάλογο που θα είναι πολύ περιγραφικός είτε να κλείνει προς οποιαδήποτε κατηγορία αδικήματος ή θύματος. Βεβαίως αυτό είναι δύσκολο από την πλευρά της Επιτροπής Γυναικών, το αντιλαμβάνομαι και πράγματι όλοι αναγνωρίζουμε πως υπάρχει μια ιδιαίτερη ευπάθεια όσον αφορά τα παιδιά. Και αυτό πρέπει να αναφερθεί στην κατάσταση των παιδιών. Αλλά αν γίνουμε πολύ περιγραφικοί, χάνουμε την η ικανότητα να δώσουμε την απαραίτητη βοήθεια στα θύματα. Οπότε ελπίζω πραγματικά να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία, να είμαστε σίγουροι πώς θα δούμε όχι μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός θύματος σε μία κατηγορία, αλλά και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε θύματος και του κάθε αδικήματος. Ε, την φύση του αδικήματος, τη φύση του εγκληματία και βεβαίως όλα τα ε, πραγματικά περιστατικά. Χρειάζονται πόροι βεβαίως για να επιτευχθεί αυτό αλλά κατά την άποψή μου μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε την βοήθεια η οποία είναι απαραίτητη και χρειάζεται νομίζω στην γενική διατύπωση αυτή και για να είναι αποδεκτή και από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ κυρία Λέτφορτ. Thank you very much. Um, ευχαριστώ. Η κυρία Κρίσπα είναι η σκιώδης. Ε, αλλά ε, θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου, διότι πρέπει να πάω πίσω στην Επιτροπή της ε, ΛΥΜΠΕ σύντομα. Συμφωνώ και υποστηρίζω ε, το έργο των εισηγητών μας στον τριμερή διάλογο που είναι μια πολύ ξεκάθαρη δουλειά ε, για μια ισχυρή οδηγία σχετικά με τα θύματα. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές νομίζω και πρέπει να υπάρξει κάποιο συμβασμό αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και νομίζω ότι στο άρθρο 7 και στο άρθρο 13, το άρθρο 7 είναι το δικαίωμα για μετάφραση και διαρμηνία και το 13 είναι για αποζημίωση των εξόδων, το θέμα των πόρων ασφαλώς προκύπτει. Και αυτό που είναι λογικά σωστό να απαιτήσει κανείς από τις χώρες μέλη να καλύψουν είναι ακριβώς αυτό. Υπήρχε μια φράση στο κείμενο του Συμβουλίου σχετικά, μια φράση που μιλούσε για τις χώρες μέλη οι οποίες διασφαλίζουν την υποστήριξη αυτή προς τα θύματα σύμφωνα με το ε, σύστημα ποινικής, ε, του ποινικού κώδικα. Εγώ βλέπω με καλό μάτι αυτή την διατύπωση. Βέβαια μπορούμε να πούμε ενεργό συμμετοχή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρξει μια διατύπωση αρκετά περιοριστική που αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ένα θύμα το οποίο λαμβάνει ενεργό μέλος, μέρος στις διαδικασίες. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα καθορίζεται αυτό που είναι υποχρεωτικό να αναλάβουν οι χώρες μέλη. Δηλαδή, να προσφέρουν ελεύθερη μετάφραση διερμηνία και αποζημίωση των δαπανών. Από την άλλη, δίδεται αγώνας για να περιοριστούν οι δαπάνες ε, και τα έξοδα σχετικά με τις δικατιστικές διαδικασίες και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν υπάρχουν πολλά λεφτά να κυκλοφορούν αυτή, στις μέρες μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει υποχρέωση έναντι του θύματος που λαμβάνει ενεργό μέλος της διαδικασίας και αυτού που δεν το πράττει διότι είναι προφανές ότι έχει δικαίωμα να το κάνει ή όχι, αλλά αν το κράτος έχει την υποχρέωση να πληρώσει και να αποζημιώσει τα θύματα, είναι ένα διαφορετικό θέμα. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο με αυτή τη διατύπωση, μάλλον ε, πιστεύω ότι μια πρόταση σύμφωνη με αυτή που είπα προηγουμένως, δηλαδή οι χώρες μέλη να προσφέρουν την απαραίτητη αρρωγή όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία τους, θα ήταν κατάλληλη σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι η έκκλησή μου, ώστε να έχουμε μια ρεαλιστική στάση ως προς το τι ζητούμε να κάνουν οι χώρες μέλη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κρίσμπεκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω αυτή την εξαιρετική πλήρη εργασία από τις δύο συντάκτριες και όπως είχα την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω την ποιότητα στις δύο επιτροπές των εργασιών, παρόλο που κάπως μπερδεύονται τα πράγματα όσον αφορά το χρόνο, το συνδυασμό, γιατί στην Επιτροπή Ελευθεριών ακριβώς είχαμε συνάντηση την ίδια ώρα σήμερα το απόγευμα, δυστυχώς, δυστυχώς και θα ήθελα πάντως ε, να χαιρετήσω την πολύ καλή δουλειά που θαυμάζομαι και να ευχαριστήσω για την αποτελεσματικότητα και να σας διαβεώσω για την πλήρη υποστήριξή μου για οτιδήποτε πρόκειται ακόμα να συμπληρωθεί, να χτενιστεί κλπ. για να φτάσουμε σε μια γοργή συμφωνία για αυτό το θέμα που όπως το υπενθυμίσετε ενδιαφέρει άμεσα πολλά εκατομμύρια πολιτών της Ευρώπης. Είναι περίπου το 15% που είναι δυνάμει θύματα και περίπου 75 εκατομμύρια δηλαδή κάτοικοι, πολίτες που αφορά το θέμα και στα πλαίσια της ρύθμισης ευρωπαϊκής εδώ πρόκειται για ένα κείμενο που ιδιαίτερα μπορεί να απασχολήσει, να ενδιαφέρει τους πολίτες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτή η ισορροπία, γιατί το να μιλάει κανείς για τα θέματα είναι πολύ σημαντικό κατά την απόψή μου και κυρίως η όλη ποινική διαδικασία και για να μπούμε στο κέντρο του προβλήματος θα ήθελα να θίξω το θέμα των άρθρων που, για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως και που αποτελούν ενδεχόμενα αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, για την υπεράσπιση το 5, 7 και 10 άρθρα τα οποία συζητήθηκαν στο τέταρτο τριμερή χθες διάλογο και να υποστηρίξω τη θέση σας ε, που θα λέμε ότι από τη στιγμή που επανασυντάσσεται η οδηγία η πανασύνταξη αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωσή της, δηλαδή με καλύτερη προστασία και όχι να πιστοχωρήσουν αυτά και να έχουμε λιγότερη προστασία και εμείς οι πράσινοι εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε με τον τρόπο αυτό και κάτι ακόμα όπως το υπενθύμησε άρρωστε, άλλωστε και η συνδάκτρία συνεισηγήτρια θα ήθελα να συγχαρώ για το ότι λαμβάνουν υπόψη, λαμβάνουν υπόψη τα παιδιά Βλέπουμε πολλές συμβαστικές προτάσεις και τροπολογίες και στο πρώτο άρθρα της οδηγίας την προσθήκη αυτή τη δυνατότητα για μία παράγραφο που να επενθυμίζει αυτή την παραπάνω ακόμα προστασία για τα παιδιά γιατί θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το συμφέρον του παιδιού και την προστασία του και θα πρέπει ίσως αυτό το πρώτο εδάφινο το επαναπεξεργαστούμε αλλά όλα αυτά προωθούνται και νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Για τη συμβαστική λύση που ιδιαίτερα σκληρά για το άρθρο 23 διαπραγματευτήκατε και εδώ για την όλη διαδικασία όσον αφορά την εγκληματική αυτή θα πρέπει να το δούμε, όπως επίσης και αυτό που υπενθυμίσετε πριν από λίγο, το ότι εξετάστε και πάλι αυτά τα πρότυπα που λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης και υποστηρίζει, αφορά το άρθρο 22, και που έχουν συμπεριληφθεί και εφαρμόζονται σε κάθε θύμα που έχει ειδικέ απαιτήσει ανάγκες και πέρα από τα ελάχιστα απαραίτητα για τα παιδιά και οι ακροάσει να λαμβάνουν χώρο για να κρίσει και λοιπά σε ειδικού χώρους και επίσης αυτή η αρχή που με απασχολούσε ιδιαίτερα για το ότι θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες στα πλαίσια αυτών των ανακρίσεων που θα ασχολούνται με την υπόθεση και ακόμα για το άρθρο 24 για τη συμβαστική λύση για την εκπαίδευση του προσωπικού κατάλληλη όπως πρέπει και όλοι έτσι έχουν επαφή με τα θύματα. Λοιπόν, αυτό αυτοί οι επαγγελματίες ειδικά εκπαιδευμένοι αυτή η ιδέα και όχι μόνο οι ειδικοί δικαστικοί αλλά οποιοδήποτε άλλο έχει επαφή με τα θύματα αυτό κατά την απόψή μου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο όπως η αστυνομία, ε, και το όλο προσωπικό σε οποιαδήποτε υπηρεσία, νομική, το να άλλο, όλα αυτά βελτιώνουν τα πράγματα όσον αφορά το προηγούμενο κείμενο. Ολοκληρώνοντας δε, η κοινοβουλευτική ομάδα θα υποστηρίξει και τα εκκρεμή σημεία όπως το άρθρο 21 για αυτή την εκτίμηση κατηγορίας την περίφημη που νομίζω ότι είναι δύσκολο σημείο, χρειάζεται να το επεξεργαστούμε αλλά επαναλαμβάνω ότι την εργασία αυτή τη θεωρώ πραγματικά ιδιαίτερα τεχνικής φύσεως δύσκολη, αλλά πάντως πλήρης ε, σχεδόν ε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, έχω το όνομά μου τώρα στον κατάλογο και θα μιλήσω σου ειδικά. Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Eh, jag kan också naturligtvis, som jag redan gjort, eh, fylla i lovsången om att... Λοιπόν, ε, και εγώ θα μπορούσα να ημενήσω ε, ενθουσιοδός την επιτυχία των ισχυριτών δεν υπάρχουν ισχυώδει συζητητές, αλλά εν πάση περιπτώσει προς όλους μπορώ να πω ότι κάνατε φανταστική δουλειά και έχει σημειωθεί και πρόοδος. Ωστόσο, υπάρχουν δύο σημεία που θα ήθελα να θίξω. Πρώτον, σχετικά με το άρθρο 8. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής παραμένουν πολύ καλύτερες. Της Επιτροπής μας εννοώ. Τώρα, αν κάνουμε τη σύγκριση ποιες προτάσεις είναι καλύτερες, ε, οι καλύτερες είναι της δικής μας Επιτροπής, οι δεύτερες καλύτερες είναι της Κομισιόν και οι τρίτες και χειρότερες είναι του Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό που έχουμε την προοπτική του φίλου καταρχήν. Ωστόσο, οι θέσεις του Κοινοβουλίου ηχούν πολύ, με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία της Επιτροπής το βλέπει αυτό. Το βλέπει κανείς και στους ορισμούς στο άρθρο 2. Το ίδιο ισχύει. Αν δηλαδή δεν υπάρχει ένας ο σωστός ορισμός της βίας με βάση τη διαφορά του φύλου, δεν θα έχουμε και πολλά αποτελέσματα. πρέπει να δώσουμε τον ορισμό αυτού που πραγματικά είναι. Και όταν κάνουμε χρήση του όρου βία επί τη βάση του φύλου, πρέπει να ξέρουμε περί τίνος ομιλούμε. Αν κοιτάξετε το παρελθόν, το ιστορικό, η Κομισιόν δεν εφλέγεται και πάρα πολύ να προωθήσει αυτή την οδηγία σχετικά με τη βία που ασκούν οι άνδρες εις βάρος των γυναικών. Αυτές οι πτυχές λοιπόν θα πρέπει να διατηρηθούν. Τώρα, ως προς τους ορισμούς, βλέπετε ότι το άρθρο 2 συγκεντρώνει τεράστια υποστήριξη στην Επιτροπή. Δηλαδή, απαιτείται ο ορισμός της βίας βάση του φύλου. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο έργο σας και ελπίζω ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο τελικά θα πιστούν και θα λάβουν υπόψη τις δικές σας θέσεις. Τόσο η Λίμπια όσο και η ε, Επιτροπή Γυναικών έχουν ε, στεναρές θέσεις επί των θεμάτων αυτών. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Πέρες. Εδώ σήμερα το πρωί εντάξει κανονικά εδώ με είπαν Πέρες αλλά το όνομά μου είναι για να τιμήσω και τη μητέρα μου Γκαρθία Πέρες τέλος πάντων να αναφερθώ στην όλη συζήτηση για τον εκπρόσωπο της Δανικής Προεδρίας θα ήθελα να πω ότι ε, οι διαπραγματεύσει από πλευρά κοινοβούλου ήταν πολύ σκληρέ αλλά και ιδιαίτερα επιδέξιε. Και οι υπόλοιποι από τι δύο επιτροπέ ε, είχαμε εμπιστοσύνη στην όλη διαπραγμάτευση. Ήταν όμω δύσκολε και παρόλα αυτά επιδέξιες. Εδώ θα πρέπει να δούμε, όπως ακριβώς είπε και ο Πρόεδρος, το θέμα ήταν σημαντικότατο για μας να ορίσουμε ποια είναι τα θύματα ε, βίας λόγω του φίλου τους και είναι πράγματα που χρειάζεται πάντα να υποστηρίζουμε. Πάντως η εργασία που έγινε ήταν πολύ καλή. Έχετε την πλήρη εμπιστοσύνη μας στην εργασία αυτή. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό σχετικά δηλαδή με την άξη βίας λόγω φύλου Χρειάζεται να το προσέξουμε αυτό, να επιμείνουμε σε αυτό, να επιμείνουμε στη θέση μας και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια συμφωνία με το Συμβούλιο ώστε να συμβαδίσουμε, να συγκλίνουμε προς το στόχο που έχουμε ρίσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε την κυρία Μπογκαρσία Πέρες, όχι Σκέτο Πέρες σαφώς θα βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο σας απευθύνω το λόγο στο άμεσο μέλλον, υπόσχομαι. Και τώρα τον τελευταίο λόγο έχουν οι εισηγητές. Ωραία. Θα αρχίσω με το πιο δύσκολο θέμα. Τη βία βάση φύλου και τη βία σε στενές στο πλαίσιο στενών σχέσεων. Και αφού το Συμβούλιο είναι παρόν εδώ, θα διαπιστώσει τις στεναρές θέσεις και των σκιωδών και πόσο αυτή η Επιτροπή επιθυμεί να υπάρξει ορισμός και να προσδιορίζονται αυτά τα ειδικά εγκλήματα. Εν τω μεταξύ σας δώσαμε και τους απαραίτητους λόγους για τους οποίους επιμένουμε οπωσδήποτε ε, σε αυτά τα σημεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι υπάρχουν κενά στις εθνικές νομοθεσίες αλλά και στις όλη διαδικασία ε, σημειώνουν, υπάρχουν σημεία αμέλειας και διακρίσεων εις βάρος των θεμάτων. Χρησιμο, καθώς χρησιμοποιούνται οι όροι αυτοί σε ολόκληρη την οδηγία, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρείτε το σωστό σημείο να βάλετε τους ορισμούς είτε στο άρθρο 2 είτε κάπου αλλού μέσα στο κείμενο σε κάποια άλλα άρθρα. Νομίζω ότι θα βρούμε μια καλή λύση αλλά αυτή είναι η στεναρή βούληση της Επιτροπής μας αλλά και του Κοινοβουλίου γενικότερα, να υπάρξουν αυτοί οι δύο ορισμοί. Στο άρθρο 7 τώρα, το οποίο ε, το εξετάζουμε ως πακέτο με το 5 και το 10. Δυστυχώς η συνάδελφος άλλη Κότφορντ δεν είναι εδώ. Κοιτάζουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις και προσπαθούμε όποτε είναι δυνατό να μην δημιουργούμε διπλά πρότυπα, διπλά στάνταρτς, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο του θύματος στην όλη διαδικασία. Δηλαδή όχι μόνο στο 5, 7 και 10, αλλά και σε άλλα άρθρα, τούτο λαμβάνεται υπόψη. Ως προς την ε, κατάρτιση, στο άρθρο 24. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα από τα λίγα κείμενα που ακόμη και το Κοινοβούλιο σημαντικά ενίσχυσε την ποιότητα του κειμένου. Δηλαδή συμφωνήσαμε σχεδόν χωρίς προβλήματα ότι απαιτείται καλή κατάρτιση και εκπαίδευση καλής ποιότητας, ούτως ώστε να γίνεται σωστή διάγνωση των αναγκών των θυμάτων και να προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες από όλες τις χώρες μέλη. Θεωρώ ότι είχαμε καλή συνεργασία από αυτού. Επίσης, σχεδιάσαμε ακόμα ένα γύρο για τον τριμερή διάλογο στις 7 Ιουνίου και πιστεύουμε ότι θα βρούμε μια καλή συμβιβαστική λύση. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες, τους συμβούλους, τους βοηθούς, τους κοιόδης και όλους όσοι δούλεψαν σε τεχνικό επίπεδο για να μας προσφέρουν συμβιβαστικά κείμενα επί των θεμάτων εκείνων που υπήρχαν αντικρουόμενες θέσεις καταρχήν. Στη συνέχεια όμως ανεβρέθη η λύση. Ελπίζω ότι και στον επόμενο γύρο θα μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε, αφού προχωρήσουμε, να οριστικοποιήσουμε αυτή την νομοθεσία και απευθύνω έκκληση, ισχυρή έκκληση προς το Συμβούλιο, παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα θέματα εκείνα που οι ευρωβουλευτές ε, θέλουν, αναζητούν λύση και να, μπορέσουν, να μπορέσει το Συμβούλιο να πείσει και τις χώρες μέλη πόσο χρήσιμο θα είναι κάτι τέτοιο να περάσει στην εθνική νομοθεσία και αυτή η νομοθεσία να εφαρμόζεται με ισότιμο τρόπο σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τις εισηγήτριες. Με συγχωρείτε. Γρήγορα, γρήγορα να προσθέσω κάτι. Η έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή μιλούσε πάντα καθαρά για το, το δικαίωμα ενημέρωσης για όλα τα θύματα ανεξάρτητα από το τι έγινε διαδικαστικά και στο Κοινοβούλιο το χαρακτήριζε πάντα το ίδιο πνεύμα και για την ε, Επιτροπή Λίμπε είναι σημαντικό. Και εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε πάνω στο σημείο αυτό μια συμφωνία. Κίπκον και Λάτφορντ, ε, οι δύο εισηγητές, ε, βλέπουμε ότι τους απασχολούν αυτά τα σημεία και μερικά κράτη-μέλη έδειξαν ε, ακριβώς ότι τα απασχολούσαν τα κράτη-μέλη για το κόστος αλλά να μην πληρώνουν τα θύματα αυτό το κόστος για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες αποτελεί ελπίδα θύματα εγκλήματος και έχουμε την υποχρέωση για αυτά τα θύματα να βελτιώσουμε την ε, στήριξή τους και να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά τους ε, και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τις κατάλληλες θέσεις και λύσεις. Το είπαμε ήδη ε, στο Συμβούλιο ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν όπως πρέπει. Αλλά για να μπορέσουμε να πετύχουμε μην αφήνουμε στην άκρη δικαιώματα που είναι αυτονόητα. Δεν θα πρέπει να τα αγνοούμε, να τα παρακάμπτουμε. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, πώς έχει όλη η διαδικασία, πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά την απόψή μας και σύμφωνα με το άρθρο 21, που όπως είπαν οι σκιώδεις ηγητές, είναι επίση σημαντικό και θα προσπαθούμε να βρούμε μια κατάλληλη λύση για να τονίσουμε ιδιαίτερα τη μορφή αυτή εγκλήματος για τα θύματα αυτά, να μην θίξουμε κανένα, να μην παραλείψουμε κάτι και θα προσπαθήσουμε όπως είπαν και άλλοι να είμαστε σκληροί και επιδέξει, εντάξει όχι αναγκαστικά σκληροί, αλλά τουλάχιστον έξυπνοι και να λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των θυμάτων και γιατί πάνω στο δικό τους το πετσί τα δοκιμάζουν αυτά και υποφέρουν και εμείς ε, οποιαδήποτε από εμά μπορεί να είναι θύμα και ακριβώς ε, μπορεί ε, να ευγνωμονεί αύριο τους συντάκτες αυτής της ρύθμισης, αυτής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες και την κυρία Χιμένεθ που συμπροέδρευσε μαζί μου. Ευχαριστώ την Επιτροπή Ελευθεριών για το ότι οργανίσαμε αυτή την ε, κοινή συνεδρίαση και άρα λύεται εδώ πέρα η συνεδρίαση η κοινή και σε ένα λεπτάκι ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μιλήσω σουηδικά από εδώ και μπρος. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Okay, we, we start... Ωραία. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, ναι. Σουηδικά. Το πρώτο θέμα λοιπόν αφορά ένα χρηματοδοτικό μέσο και την σύσταση του. Δυστυχώς κυρία Ματέρα δεν είναι εδώ σήμερα. Οπότε έχει μια πρόταση. Ξέρω πως η κυρία Μπαστός θα την αντικαταστήσει. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η, δυστυχώς η συγγήτρια Μπάρμαρ Ματέρα είναι απούσα σήμερα και μου ζήτησε μέσω ενός σημειώματος να το διαβάσω εδώ. Το Δεκέμβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο ένα κανονισμό για ένα εργαλείο χρηματοδότησης ε, για περισσότερη δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο στην παγκόσμιο σκηνικό. Εμείς παίζουμε σημαντικό ρόλο για την πρόσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το άρθρο 2 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί αξίες όπως την αξινοπρέπεια, τη δημοκρατία, την ισότητα και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί πολλά μέσα εργαλεία οικονομικής συνεργασίας και τεχνικής συνεργασίας για οικονομική συνεργασία σε τρίτες χώρε Εδώ προβλέπονται όμω προϋποθέσεις, κριτήρια δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να είναι σημαντική συνιστόσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα δικαιώματα της γυναίκας εδώ η συγγήτρια έχει συμπεριλάβει, παρουσιάζει τροπολογίες με σημαντικά σημεία για τη συμμετοχή στην όλη διαδικασία της γυναίκας και μια σχέση ανάμεσα στην ισότητα των φύλων και στην προστασία της δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι κοπέλες και οι γυναίκες γενικά πολλές φορές είναι τα πρώτα θύματα είτε όταν έχουμε μια μετάβαση προς τη δημοκρατία και εδώ δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου σε πολλές από αυτές τις χώρες, είτε υποεκπροσωπούνται στον, στα κοινοβουλιά τους εδώ στην όλη διαδικασία τη δημοκρατική δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς μια κατάλληλη συμμετοχή των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις διάφορες δύσκολες καταστάσεις όπως με στρατιωτικά πραξικοπήματα είτε φυσικές καταστροφές όπου βλέπουμε ότι ακόμη περισσότερο δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη δεύτερη τροπολογία η συνάδελφο Μπατέρα τη ζητάει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βία κατά γυναικών κοριτσιών σε περιπτώσεις ένοπλης σύραξης. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ότι υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, έκτακτες συνθήκες και είναι ακόμα πιο ευάλωτες οι γυναίκες Τροπολογία 3. Η συνάλφο τονίζει τη σημαντική αυτή πτυχή της συμμετοχής γυναικών στην πολιτική ζωή και το πώς μπορούν να ψηφίζουν, πώς μπορούν να είναι ίδιες υποψήφιες στις εκλογές. Χωρίς μια εκπροσώπηση κατάλληλη των γυναικών, η όλη δημοκρατική διαδικασία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν δημοκρατική. Διαφορετικά ένα από τα δύο φύλλα θα υποεκπροσωπείται. Και επίση η γήτρια τονίζει ότι οι αντιπροσωπείες για μια, ένα έλεγχο της προεκλογικής εκστρατείας και της ψηφοφορία των εκλογών θα πρέπει οι αντιπροσωπείε αυτέ να αποτελούνται από ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών. Έτσι, περισσότερη ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή ακριβώ των γυναικών στην πολιτική ζωή μια χώρας. Επίση, η συγγήτρια θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πάνω στο soft power να επιμείνει, δηλαδή να υπάρξουν διάφορες προϋποθέσεις πριν να δώσει κονδύλια για τη στήριξη τρίτων χωρών. Αυτή η αρχή νομίζουμε ότι λειτουργεί σωστά και έτσι οι αρκετές χώρες μπορούν να έχουν απτές βελτιώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βοηθήσει για την εξωτοποίηση των γυναικών, για τη χειραφέτησή τους παντού και σε διάφορους τομείς. Επίσης, η συνάλφος περιμένει τις εκτιμήσεις της δικές μας και τις ενδεχόμενες τροπολογίες της περιλάβει στην εργασία της. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Νεβεντάλοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Είμαι σκιώδη συγκητρία για τους ε, σοσιαλιστές. Θεωρώ πως αυτό το οποίο προτάθηκε είναι πολύ θετικό και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Έχω μόνο μία πρόταση εκεί πέρα που λέει πως ε, τα ψηφοδέλτια πρέπει να ε, περιέχουν ε, αλλά και οι αποστολές παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαρτίζονται από ίσο αριθμό άνδρων και γυναικών. Να πάω παραπέρα. Όταν νέες χώρες εκδημοκρατίζονται, να επιμένουμε πάντα να συζητηθεί το θέμα της ισότητας των γυναικών, κάτι το οποίο πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε συζήτηση όπου εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Κοινοβούλιο σε τρίτες χώρες ε, η συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει πάντα να υπάρχει αυτή είναι η τροποποίηση που έχουμε προτείνω με όλα τα άλλα συμφωνώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος τον λόγο η Κομισιόν λοιπόν ήθελε να παρέμβει όχι. Αν μου επιτρέπετε, είμαι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, μέλος της ομάδας ε, που διαπραγματεύεται το Ευρωπαϊκό Μέσο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βεβαίω η Κομισιόν ε, είναι επικεφαλής. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω πως η διάσταση του φίλου είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του κανονισμού, πως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν. Η νέα πρόταση που είναι τώρα επιτάπητος ε, βασίζεται στην προηγούμενη πρόταση και προχωρεί παραπέρα. Αυτό το οποίο έχετε μπροστά σας, η πρόταση της Κομισιόν είναι μια εξέλιξη περισσότερο παρά μια ε, επανάσταση. Οπότε βασιζόμαστε σε αυτόν τον κανονισμό και αυξάνουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτό το μέσο διατηρώντας πάντα τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, το βάρος που δίνεται στην κοινωνία των πολιτών, στην ισότητα των φύλων, αυτά υπάρχουν ήδη στην πρόταση υπάρχει ένα εκτιμώντας ήδη μια αιτιολογική σκέψη για το ζήτημα του φύλου. Και βεβαίως ε, ένα σχόλιο για τις αποστολές παρατήρησης των εκλογών. Προσπαθούμε πάντα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει, ε, να υπάρχει η εκπροσώπηση των γυναικών, αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είτε μιλάμε για ισορροπία γεωγραφική, έχουμε και εταίρους επίσης, είτε μιλάμε ε, από την Ελβετία, από τον Καναδά και βεβαίω και τους υποψηφίους που προτείνονται και τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία προτείνουν υποψηφίους. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία και μπορείτε να βρείτε αποστολές με σημαντικό αριθμό γυναικών. Τέλος, συμφωνώ με το τελεσχόλιο σχόλιο για την διάσταση του φύλου στις αποστολές παρατήρησης εκλογών γιατί προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανάλυση και τη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Όλες οι εκθέσεις από τις αποστολές της Ένωσης περιέχουν τώρα, περιέχουν τώρα μια τέτοια διάσταση. συμμετοχή γυναικών, το εκλέγει και εκλέγεστε. Έχουμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έχουμε μια τέτοια αποστολή παρατήρησης εκλογών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο, την κυρία Παδοπουλού. Θεωρώ ότι η κυρία Ματέρα έχει κάνει πολύ καλές εισηγήσει. Στέκομαι ακριβώς στην εισήγηση που έχει κάνει ότι πρέπει οι παρατηρητέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκλογικέ αναμετρήσει πρέπει να αποτελούνται από ίσον αριθμό γυναικών και ανδρών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ακριβώ ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών. Θα σταθώ ιδιαίτερα όμως σε μια ανησύγηση που έχει κάνει ότι οι στόχοι για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ισότητα των φύλων πρέπει να εντάσσονται συνεχώς σε κάθε μέσο χρηματοδότησης της εξωτερικής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες. Εγώ θα ήθελα ακριβώς αυτή η αναφορά για την ισότητα των φύλων και για ενδυνάμωση των γυναικών να γίνεται και σε ό,τι αφορά την προενταξιακή βοήθεια που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη τώρα που η Τουρκία χτυπά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα η διάσταση του φύλου να είναι μια από τις παραμέτρους βάσει της οποίας θα αξιολογείται η πρόοδος που σημειώνει η Τουρκία σαν χώρα υποένταξη, γιατί ακριβώς εκεί βλέπουμε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και η ισότητα των φύλων δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως. Επομένως, αυτή η εισήγηση που γίνεται σε κάθε μέσο χρηματοδότησης εξωτερικής βοήθειας προς τρίτες χώρες, κατά παράλληλων τρόπων πρέπει να υπάρχει αυτή η ισότητα και να ενσωματώνεται η διάσταση των φύλων και στην προενταξιακή βοήθεια προς χώρες ε, στην ενταξιακή του διαδικασία. Και αυτή είναι η τροπολογία που θα κάνω προσωπικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν η κυρία Μπέστος ε, θα ήθελε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις ακόμα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλά και μόνο για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και τον εκπρόσωπο εξωτερικής δράσης εξ ονόματος της εισηγήτριας να σας πω ότι σημείωσα όλα αυτά τα σχόλια και θα τις επιταβιβάσω τα όσα άκουσα σήμερα εδώ, τα διάφορα σχόλιά σας για την έκθεσή σας. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίδραση, το αντίθετο, συμφωνείτε μάλλον. Σας ευχαριστώ. Τελειώνουμε με αυτό το σημείο. Να σας πω πως η προθεσμία και τροπολογίε είναι 4 Ιουνίου, 5 ώρα το απόγευμα και η Επιτροπή μας θα ψηφίσει στις 21 Ιουνίου. Η Επιτροπή Εξωτερικών θα ψηφίσει στις 10 Ιουλίου. Και τελειώσαμε με αυτό το θέμα, περνάμε στο επόμενο. Μπορεί ίσω να δούμε και το σημείο 20 τη ημερήσια διάταξη. Βεβαίω, 5 λεπτά έχουν μείνει μόνο για τη λήξη της ε, συνεδρίασης, αλλά να αναφέρω πως είχαμε μια επίσκεψη αντιπροσωπεία στην Κύπρο. Είχα πάει με τις κυρίες Ζαμπόρσκα και Ζούπερ και Παπαδοπούλου και Θεοχάρους. Πήγαμε λοιπόν όλοι στην Κύπρο θέλαμε να επισκεφτούμε την Κύπρο πριν από την Κυπριακή Προεδρία. Είχαμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, πολλές συναντήσεις, νομίζω πως θα δείτε τις πληροφορίες στο έγγραφο που έχετε. Έχουμε πάρα πολύ καλές επαφέ Να πω συνοπτικά πως έχουμε την εντύπωση πως η Κυπριακή Προεδρία Προεδρία θέλει να διασφαλίσει πως αυτά τα ζητήματα θα είναι υψηλά στη ημερήσια διάταξη. Και βεβαίως έχουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο που εργάζονται σε αυτά τα ζητήματα ε, και θέλουν να τα προωθήσουν. είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες επαφές με την κυβέρνηση, ΜΚΟ κτλ. και βουλευτές. Ίσως να μου πω τίποτα άλλο, κυρία Λούμπε. Ah. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι κατά την άποψή μου η επίσκεψη αυτή ήταν μάλλον θετική λόγω των επαφών ε, που είχαμε, λόγω της οργάνωσης δεν ήταν μόνο θεσμικής κυβερνητικής φύσεως, ούτε και κοινοβουλευτικής, ε, παρόλο που ήταν συνάδελφοι παρόντες και βουλευτές ε, και στελέχη κυβερνητικά. Χάρηκα όμως που δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για να έχουμε σχέσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλες ενώσεις που εργάζονται εκεί και ασχολούνται άμεσα με θέματα γυναικών και ισότητας των φύλων. Και ακούσαμε και το τι έχουν αποκομίσει σαν εμπειρίες επιτόπου τις εντυπώσεις τους και νομίζω ότι όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμα για να έχουμε μια ακριβή ιδέα για το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Πέρα από αυτά που ήδη ανέφερε ο Πρόεδρος, θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με τα δικαιώματα της γυναίκας και το όλο πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα για το οποίο είχαμε συζητήσει στην ε, κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Νομίζω ότι η υποδοχή από την μελλοντική Προεδρία του Συμβουλίου ήταν ιδιαίτερα θετική και πάνω σε σημεία που ιδιαίτερα μας απασχολούσαν όπως για τη μητρική άδεια, την οδηγία αυτή και το gender pay gap, ακριβώς τη διαφορά αμοιβή για την ίδια εργασία. Όλα αυτά εξετάστηκαν, η Κυπριακή κυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερα σημασία σε αυτά. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να προσχεδιάζουμε εν ώψη της Κυπριακής Προεδρίας. Ακόμα μερικές ειδικότερες ε, θέσεις ε, που αφορούν την Κύπρο. Δηλαδή, την ειδικό χαρακτήρα της γυναίκας ε, στην Κύπρο. Εμείς ανησυχούσαμε για μερικά πράγματα. Ακούσαμε όμως απόψεις από διάφορες οργανώσεις και από κυβερνητικά στελέχη. Εδώ ας πούμε για το εμπόριο κατά πούμε γυναικών, μάλλον την παράνομη μετανάστευση πολλών γυναικών που φτάνουν στην Κύπρο και μετά εργάζονται κάτω από από δυσμενείς, ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες χωρίς να απολαμβάνουν κανένα δικαίωμα. Απολύτως κανένα. Αυτό όμως δείχνει ανάγλυφα αυτό το πρόβλημα της εκμετάλλευσης των γυναικών, του παράνομου αυτού εμπορίου, τόσο απέσιο αυτό το παράνομο εμπόριο που δεν έχει όμως ξεπεραστεί ούτε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν εκ νέου. Και ακόμη κάτι. Μιλήσαμε για την πολιτική ισότητα φύλων στην Κύπρο. Όπως επίσης για διάφορες δράσεις σε εθνικό επίπεδο. Είναι αρκετά προχωρημένη η νομοθεσία, πάνω για την βία κατά των γυναικών. Τώρα από την νομοθεσία μέχρι την πραγματική αντιμετώπιση εκεί διάφορες δυσκολίες. Η νομοθεσία καλή, μάλλον καλή είναι. Απαιτείται όμως μια εργασία το πώς όλα αυτά θα εφαρμόζονται πραγματικά γιατί στην καθημερινή πρακτική υπάρχουν δυσκολίες. Επίσης να θίξω κάτι που με απασχόλησε προσωπικά, μου έκανε εντύπωση. Ήταν η πρώτη μου φορά που πήγαινα στην Κύπρο με εξέπληξε γιατί είδα ότι εντάξει αυτό θα εξέπλησε σε οποιαδήποτε χώρα αλλά σε μια χώρα ε, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα δικαιώματα των πολιτών της καθημερινά παραβιάζονται επειδή εκεί επεμβαίνει μια άλλη χώρα που σχεδόν τη μισή χώρα κατέχει αυτό όχι μόνο με εκπλήσει αλλά με σοκάρει είναι μια κατάσταση που παρατηρείται από το 1974. Και ακόμα περισσότερο μας σοκάρει εδώ. Πολύ συχνά μιλάμε για διεθνή συνεργασία, για προώθηση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μερικές φορές, όμως όλα αυτά είναι αρκετά αφηρημένα, είναι αρκετά μακριά από την καθημερινή ζωή. Εν έχουμε δίπλα μας παραβιάσεις, ε, απέσια σχήμες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να εφαρμοστούν και οι αποφάσεις των Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζονται τα δικαιώματα του κυπριακού λαού που υφίσταται την κατοχή ενός τμήματος της χώρας και την απομάκρυση πολιτών από εκεί που γεννήθηκαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε ο χρόνος μας. Θα περάσουμε συνεδρία στον συντονιστών. Ε, πρώτα απ' όλα θα μιλήσει η κυρία Παπαδοπούλου για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να πω ότι ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση που είχαμε ω αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήμουν ιδιαίτερα ευτυχή να συναντήσω συναδέλφου ε, που ήρθαν στην Κύπρο. Πράγματι, στην Κύπρο πρέπει να είσαι παρόν για να αγγίξει τον τύπο των ύλων και να καταλάβει τι σημαίνει να ζει σε μια ανημικατεχόμενη πατρίδα. Η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει σαν στόχο να ασχοληθεί με ευρωπαϊκά θέματα ε, και ένα από του στόχου είναι από πλευρά του του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναδείξει ακριβώς την πτυχή της βίας κατά των γυναικών. Θα γίνουν ε, μεγάλες συναντήσεις και εκδηλώσεις και στην Κύπρο και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της βίας. Ε, θα πρέπει να πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1984 εφάρμοσε μια πολύ προοδευτική νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που αποτελούσε μια καλή πρακτική και το είχαμε σχολιάσει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σίγουρα η νομοθεσία είναι εναρμονισμένη όσον αφορά τα θέματα ισότητας των φύλων, αλλά στην εφαρμογή πάντα υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα. Ε, είχαμε την ευκαιρία ε, με την Επιτροπή ΦΑΜ, την Αντιπροσωπεία, να συζητήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, το μισθολογικό χάσμα. Είναι γεγονό ότι και στην Κύπρο το ποσοστό γυναικών στη Βουλή εξακολουθεί να είναι χαμηλό, ενώ τελευταία είδαμε πρόοδου όσον όσον αφορά το διορισμό γυναικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε ψηλέ θέσει στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Αλλά ακόμη έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Και να πω ότι ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί είναι η ενσωμάτωση των ε, γυναικών που είναι μετανάστριες και εργάζονται στον τόπο μας ως οικιακέ βοηθοί και ο στόχο είναι ακριβώς να ενσωματωθούν στην κυπριακή κοινωνία όπω ε, όπως ε, και εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, να πω ότι εμεί καλωσορίζουμε κάθε επίσκεψη από Ευρωπαίου συναδέλφου, γιατί είναι μια ευκαιρία ακριβώ να δουν και τη σημαία των πενταδάχτυλων. Υπάρχει μια τουρκική σημαία χαραγμένη πάνω στην οροσυρά του πενταδάχτυλου και όσοι ξένοι έρθουν εκεί και τη δουν πραγματικά σοκάρονται γιατί πολλέ φορέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλούμε για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτε χώρε, αλλά στη δική μου πατρίδα στην Κύπρο όσοι επισκεφτούν θα δουν ότι τέτοιε παραβιάσει συνεχίζονται τα τελευταία 38 χρόνια από την κατοχική Τουρκία. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα. Έχουμε συντάξει την έκθεση σχετικά με την επίσκεψη αυτή. Έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε την έκθεση με την άνεσή σας. Σημείο 21, τα διάφορα, δεν υπάρχουν άλλα διάφορα. Σημείο 22, προσεχή συνεδρίαση. Η προσεχή θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου από 3 έως 6.30. Και επίσης θα έχουμε και μια ακρόαση για την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική. τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η λήξη αυτής της συνεδρίασης και σε 30 δευτερόλεπτα θα επιστρέψουμε για τη συνεδρίαση των συντονιστών.